La séance est ouverte. Le commissaire est dans nos murs. Il nous rejoint dans quelques instants. Άρχεται η συνεδρίαση. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ε, και ο Επίτροπος. Ε, να σας πω ότι τα σημεία της Μέσης διάταξης έχουν τροποποιηθεί η σειρά τους, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα υπάρξει ψηφοφορία για τα σημεία 3, 4 και 5 του προπολογισμού 2019. Τμήμα 3 ε, Επιτροπή και άλλα τμήματα καθώς και η πολιτική ε, για τα κτίρια θα το δούμε μετά το σημείο 7. Το 345 μετά το 7. Ενώ το σημείο 8 θα το δούμε πριν το σημείο 7. Το σημείο 8 είναι για τον Brexit. Προσανατολισμό ε, ε, για τον προπολογισμό του 2020. Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση, τροποποιείτε λοιπόν η διάταξη όπω μόλι σα ανέφερα. Να σα πω επίση ότι οι αποφάσει των συντονιστών που πάρθηκαν στι 23 Ιανουαρίου περιλαμβάνονται στο φάκελο της συνεδρίασης. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, ε, μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Μια πράξη κατεξιοδότηση μας κοινοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2018. Λάβαμε λοιπόν την εξής πράξη κατεξιοδότηση της Επιτροπής στις 18 Δεκεμβρίου του 2018 που αφορά τον, τον, τον οικονομικό οργανισμό πλαίσιο για του οργανισμού που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη Ευρατόμ και αφορά το άρθρο 70 του κανονισμού 2018. 846 ε, ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Έχουν δύο μήνες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στη διάθεσή τους. Ε, μπορεί να υπάρξει μια παράταση ακόμα δύο μηνών για να ε, εκφράσουν οποιαδήποτε αντίθεση σε αυτή την πράξη κατεξουδότηση. Σύμφωνα με μια γραπτή διαδικασία, οι συντονιστέ τη Επιτροπή Προπολογισμού και τη Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου αποφάσισαν να μην παρατείνουν αυτή την προθεσμία και να μην διταχθούν στην πράξη κατεξουδότηση. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, η απόφαση αυτή ε, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Το Συμβούλιο ζήτησε παράταση της προθεσμίας για δύο μήνες ε, και βεβαίως καλωσορίζω και τον επίστροπο Έτιγκερ που μόλις έφτασε για τον Brexit τώρα και πριν δώσω το λόγο στον επίτροπο που θα αναφερθεί σε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη ε, πλέον πιθανή μη συμφωνία ε, μετά από μια γραπτή διαδικασία μεταξύ των συντονιστών τη Δημοσιονομική Επιτροπή είμαι πλέον εισηγητή για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τα επίγοντα μέτρα σχετικά με την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση του προπολογισμού ε, την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του προπολογισμού 2019 που θα μα παρουσιάσει ο Επίτροπος Έτιγκερ. Η έκθεση την οποία θα προετοιμάσω θα υποβληθεί στην Επιτροπή στις 7 Μαρτίου, θα ψηφίσουμε 18 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και η Ολομέλεια πιθανότατα 8 Απριλίου θα ψηφίσει στην πρώτη λοιπόν ε, Ολομέλεια του Απριλίου αυτά ήθελα να σας ε, ε, γνωστοποιήσω σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ μαζί μας για να μας παρουσιάσετε αυτήν την πρόταση κανονισμού θα ήθελα να θυμίσω ότι η έξοδος του Ηνωμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία Βεβαίω, βεβαίως ε, η κυρία Μέη έρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες, αλλά αυτή η έξοδος ε, αυτή τη στιγμή φαίνεται να οδηγείται να φαίνεται να οδηγούμαστε σε μια έξοδο χωρίς συμφωνία και θα πρέπει επίτροπος να μας μιλήσει για τα μέτρα που θα να παρθούν σε σχέση με το δημοσιονομικό αντίκτυπο για τον προπολισμό του 2019 αλλά και τον προπολισμό του 2020. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας για να μας διαφωτίσετε. Παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Αρτουή, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω μαζί σας για, μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταθέτουμε στα πλαίσια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πρόεδρος μου ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η συμφωνία αποχώρησης είναι και εξακολουθεί να είναι η καλύτερη και η μόνη δυνατή συμφωνία. χαιρετίζουμε το γεγονό ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί μεν λύση, αλλά πάντως στο Βρετανικό Κοινοβούλιο διαμορφώνεται σαφής πλειοψηφία υπέρ ενός σενάριου με συμφωνία. Δηλαδή η πλειοψηφία επιθυμεί να αποφύγει οποιοδήποτε σενάριο χωρίς συμφωνία. Και έχουμε την ευκαιρία στη βάση του σχεδίου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αποχώρησης για να αποφευθούν μεγαλύτερες ζημιές και που φαίνεται πως ε, εγκρίνεται ε, αυτό το σχέδιο, μάλλον έχει πιθανότητα να εγκριθεί στην Βουλή των Κοινοτήτων. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον τι θα παρουσιάσει η Βρετανίδα Πρωθυπουργό σήμερα στον πρόεδρο Γιούνκερ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενη έκβαση. Θα ήταν αμελές εάν δεν είχαμε σχέδιο, το λεγόμενο contingency, δηλαδή σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή απρόβλεπτων αναγκών. Αυτή, αυτή η απρόβλεπτη η έκτακτη ανάγκη Brexit έγινε δεκτή από την Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα με βάση δική μου πρόταση. Εκ προτείνουμε ρυθμίσεις για το έρασμο συν, για τους νέους και νέες που προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στις 27 υπόλοιπες χώρες μέλη και το αντίθετο από τις άλλες χώρες μέλη δηλαδή που ε, βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορέσουν να συνεχίσουν συντεταγμένα την παραμονή τους εκεί ακόμη και μετά την ημερομηνία της 29ης Τρίτου. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση, το ίδιο, έχουμε καταθέσει προτάσεις, στη, μάλλον έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ερχόμαστε τώρα και να αντιμετωπίσουμε και το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μας ζήτησε να εντατικοποιήσουμε τις προετοιμασίες αυτές. Και το σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων του Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί άλλη μια βάση για να αντιμετωπίσουμε το αίτημα αυτό του Συμβουλίου. Προβλέπουμε μέτρα για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2019 που εγκρίνατε τέλη του 2018 εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρόκειται για μέτρα για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, δηλαδή το λεγόμενο no deal Brexit. Η πρόταση έχει χρονικό περιορισμό και περιορισμένο εύρος και εγκρίνεται μονομερός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφής εγκριθεί πρόκειται για προσφορά που κάνουμε στους Βρετανούς φίλους μας. Εάν θέλει να, ε, χρησιμοποιήσει την πρόταση αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δεχθεί ένα πλαίσιο και να το τηρήσει και υπορισμένους όρους. Μετά από την αποχώρηση το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα. Επομένως δεν εφαρμόζονται πλέον το ευρωπαϊκό δίκαιο και συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει για τις δημοσιονομικές σχέσει, δηλαδή προπολογισμού, ένα νομικό κενό. Ως συνέπεια, θεσμοί, οντότητες, φορεί που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν έδρα εκεί, δεν πρόκειται να χρηματοδοτούνται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξαίρεση έναν περιορισμένο αριθμό λίγων προγραμμάτων. Σε περίπτωση μη συντεταγμένη άτακτη αποχώρηση, δεν θα υπάρχουν πλέον νομικέ ρυθμίσει για τι δημοσιονομικέ σχέσει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 υπολοιπωμένων χωρών μελών. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά και να ρυθμιστούν εκ νέου τα πράγματα αυτά. Αυτό το νομικό κενό θα προκαλέσει σημαντική ανασφάλεια και προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού μας. Για όλους τους Βρετανούς δικαιούχου και σε πολλές περιπτώσεις και για δικαιούχου στις υπόλοιπε 27 χώρε μέλη. Ο κανονισμός που προτείνουμε έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει σοβαρές ανομαλίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 και να επιτρέψει στους δικαιούχους σε όλους τους τομείς πολιτικής, έρευνα, καινοτομία, γεωργία, να συμβάλλει ώστε να αποφευθούν προβλήματα ή πάντως να απαλληλθούν. Σύμφωνα με τον κανονισμό που προτείνουμε, θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορούσαν οι Βρετανικοί θεσμοί υπό δύο όρους να συνεχίσουν να λαμβάνουν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρώτος όρο, το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλει την συνεισφορά του για τον προϋπολογισμό 2019. Δεύτερος όρο, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Άρα ισχύουν οι ρυθμίσει για οικονομικούς ελέγχους στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η πρότασή μας περιορίζεται στο έτος 2019 χρονικά και η δυνατότητα ενισχύσεων παραμένει μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Ο κανονισμός ισχύει μέχρι τέλους του 2019 και στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για αυτήν την διάρκεια ή σχετικά με αποφάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί με αυτό το χρονικό ορίζοντα. Η πρότασή μας θα επιτρέψει και άλλες δημοσιονομικές ρυθμίσεις στο μέλλον για μια κατευθυνόμενη μετάβαση στο επόμενο έτος. Ξαναλέω τους συγκεκριμένους όρους που έχουμε προτείνει. Το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει μέχρι τις 18 Τετάρτου να έχει δηλώσει ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Θα καταβάλει τη συνεισφορά του δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2019 όπως τον εγκρίνατε και μάλιστα πλήρως. Η προθεσμία 18 Τετάρτου εγκρίθηκε ε, λαμβάνοντας υπόψη και το τέλος της δικής σας κοινοβουλευτικής θητείας. Έτσι θα μπορέσουμε στην τελευταία περίοδο συνόδου του Στρασβούργου να σας αναφέρουμε σχετικά. Μέχρι τις 18 Απριλίου θα πρέπει λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο πέραν αυτού να έχει αναλάβει την υποχρέωση να δεχθεί τους αναγκαίους ελέγχους, οικονομικούς ελέγχους, audit για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και μετά από την ημερομηνία αποχώρησή του, εάν διαπιστωθούν εκεί σημαντικές ελλείψεις, το Συμβούλιο θα μα η Επιτροπή θα μπορεί να εκδώσει απόφαση διακοπή των χρηματοδοτήσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρότασή μα είναι πλήρω αυτόνομη. Δεν αγγίζει τις δημοσιονομικές ρυθμίσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση σεναρίου χωρίς σε περίπτωση σεναρίου χωρίς συμφωνία, δηλαδή χωρίς συμφωνία. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο τηρούν τις υποχρεώσεις τους από το σύνολο των πλαισίων ρυθμίσεων που ισχύουν. Ακόμα και αν δεν έχει δηλαδή υπογραφεί η συμφωνία αποχώρησης μέχρι την 29η Τρίτου, δεν θίγονται οι ρυθμίσεις αυτές. Εμείς θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό κάνουμε μια σημαντική προσφορά για μια συντεταγμένη συνέχιση των προγραμμάτων μας που συμφέρει και τους Βρετανούς εταίρους μας θα πρέπει να αναμείνουμε τώρα να δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο, καθώ επίση και ποια θα είναι η αντίδραση των Βρετανών φίλων μα για την πρότασή μα αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση που μας κάνατε σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα δημοσιονομικά, εάν παρελπίδα δεν ε, υπάρξει συμφωνία στις 29 Μαρτίου του 19. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εισηγητές και θα με συγχωρήσετε. Ναι, ναι, όλοι θα μιλήσετε. Donc, euh, le rapporteur que je... Έλεγα λοιπόν ότι ε, οι συντονιστές και βάσει της ε, γραπτής διαδικασίας ε, έγινα εγώ ο ίδιος εισηγητής. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πάρω πρώτα εγώ το λόγο. Ε, επομένως, ε, ναι, πρέπει να υπάρξει μια δημοσιονομική ε, συνέχεια όσον αφορά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και των ατόμων ή οντοτήτων που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να υπάρξει, λέω, μια συνέχεια όσον αφορά τη συμμετοχή στα προγράμματα. Υπάρχει όμως μια, υπάρχει κίνδυνος μήπως να δημιουργηθεί μια μεταβατική κατάσταση ακόμα και σε περίπτωση μη συμφωνίας. Δεύτερη ερώτηση. Ο κανονισμός ρυθμίζει την κατάσταση της τρέχουσας χρονιάς. Τι θα συμβεί με την επόμενη χρονιά 2020. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία του προϋπολογισμού 2020. Η γενική μας εισηγήτρια Μόνικα Χαλμάγερ ήδη εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό. Τι γίνεται ε, με τα, τους ε, Βρετανούς ή τις οντότητες που ε, είναι εγκατεστημένοι τις ε, χώρες τις υπόλοιπες, αλλά έχουν σχέσεις ή δραστηριότητες συνδεδεμένες με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δε τρίτον, από ό,τι έμαθα η Κομισιόν προετοιμάζει οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που εντός του Συμβουλίου υπέβαλαν τα κράτη-μέλη. Μπορείτε να δεσμευτείτε, κυρία Επίτροπε, ότι θα δώσετε στο Κοινοβούλιο τις απαντήσεις που θα δώσετε στο Συμβούλιο και πιο γενικά κάνω μια έκκληση στην Κομισιόν να δράσει με πλήρη διαφάνεια σε σχέση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για οποιοδήποτε δημοσιονομικό θέμα σχετίζεται με την αποχώρηση χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον ερώτηση όσον αφορά δραστηριότητες ή δράσεις για τις οποίες ε, οι δικαιούχοι πρέπει να, είναι, να έχουν έναν ελάχιστο αριθμό και να προέρχονται από συγκεκριμένες ελάχιστε, από ελάχιστο αριθμό χωρών ε, στα πλαίσια μια συμπραξία ενό κονσόρσιου. Τι θα γίνει με ένα άτομο ή μια οντότητα μέλος αυτού του κονσόρσιου τη συμπράξεως που θα βρίσκεται ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι θα γίνει με τις προϋποθέσεις πληρωμής από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχω την εντύπωση ότι ε, τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν αυτό το, αυτή η σύμπραξη ε, προϋποθέτει πολλές χώρες, αλλά και μια βρετανική ε, οντότητα θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια στο σύνολο των εμπλεκομένων και να μην συνεχιστεί η καταβολή των πληρωμών. Είναι δυνατόν να προστατευτούν οι μη Βρετανοί σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μια τελευταία ερώτηση η πρόταση αποκλείει τη συμμετοχή ε, σε ε, δημόσιους διαγωνισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου άτομα, ε, αποκλείει άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν αναφέρεται ότι για λόγου ασφάλεια, ε, κάποιοι έχουν ε, άτομα ή οντότητε εγκατασταθεί σε άλλε χώρε. Αυτή είναι ιδιαίτερα ασαφή διατύπωση. μήπω μπορείτε να την ξεκαθαρίσετε κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω λοιπόν να απαντήσετε σε αυτές τις πολλές ερωτήσεις μου. Και μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές, καθώς επίσης και σε όλους όσοι εκ των συναδέλφων ε, επιθυμούν να υποβάλουν ερώτημα στον Επίτροπο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, πράγματι αυτό το σχέδιο αντιμετώπισης ε, απρόβλεπτων καταστάσεων, τέλος πάντων contingency plan, αναφέρεται πραγματικά στην περίπτωση όπου οι Βρετανοί θα αποχωρήσουν χωρίς συμφωνία. Κατά βάση δηλαδή, για να αποφύγουμε μια άμεση κάθετη πτώση. Να μπορέσει δηλαδή το αεροσκάφο να συνεχίσει να πετά και το υπόλοιπο του έτου και να προσγειωθεί ομαλά στο τέλο του. Γι' αυτό μιλήσαμε για τον Ερασμοσύν, για του ε, γεωργού, αγρότε, Ήπεθρο. Αν καταβάλουν την συνεισφορά του οι Βρετανοί, συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα τα οποία ενδιαφέρουν φορείς και πολίτες τους. Πώς θα αντιδράσουν οι Βρετανοί θα το δούμε. Το πλεονέκτημα είναι ότι θα αποφευθούν χαόδεις εξελίξεις μετά από τις 29 ε, Τρίτου και επειδή είναι καθαρή συνεισφορής οι Βρετανοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να συμβάλλουν, να, καταθέσουν, να καταβάλουν τη συνεισφορά τους δηλαδή ή όχι. Και έχουμε επίτηδες περιορίσει την ισχύ του κανονισμού στο 2019 μου ε, θέσατε έναν αριθμό ερωτήσεων. Στην ομάδα εργασίας του άρθρου 50 στο Συμβούλιο έχουμε λάβει έναν αριθμό προφορικών ερωτήσεων. Ευχαρίστως θα απαντήσουμε και στις δικές σας ερωτήσεις και στις ερωτήσεις της ομάδας εργασίας ε, άρθρου 50 εντός τριημέρου. Θα απαντήσουμε γραπτός, πλήρως, μέσα στις επόμενες Τρίτη ημέρες. Άρα το αργότερο τρίτη ή τετάρτη της επόμενης εβδομάδας θα τις έχετε. Είμαι διατεθειμένος άλλωστε ανα πάσα στιγμή να συνεχίσω και με οποιαδήποτε μορφή τον διάλογο μαζί σας. Δεν πήραμε ελαφρά υπόψη την υπόθεση αυτή. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εμείς θέλουμε να αποφύγουμε με κάθε τρόπο ένα hard crash, μια απότομη ανεξέλεγκτη πτώση. Γι' αυτό λοιπόν η ρύθμιση που προτείνουμε, ακόμα και αν δεν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης, περιορίζεται σε ένα χρόνο, σε προγράμματα του προϋπολογισμού, ώστε να αποφευθούν ζημιές εκατέρωθεν. Να μειωθούν ή, αν είναι δυνατόν, και να αποφευθούν εντελώς. Πρόεδρος Αουτουή. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. καλώντας τους ε, στο μέτρο του δυνατού να μην υπερβούν τα δύο λεπτά. Και το παράδειγμα είμαι βέβαιος θα δώσει ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω όμως πορτογαλικά. Um e Ευχαριστώ πολύ. Γενικώ είμαι αισιόδοξη ε, και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, ε, τα πράγματα θα είναι άσχημα και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω καλύτερα είναι να προλαμβάνει κανείς και όχι ε, να πρέπει μετά να θεραπεύσει, όπως λέμε και εμεί στην Πορτογαλία. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα τα ε, ερωτήματα έχουν, τα σημαντικά έχουν ε, υποβληθεί από, και από τον Πρόεδρο. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Λαμβάνοντας υπόψη τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 οι πληρωμές γίνονται την επόμενη χρονιά. Πράγμα που σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εκπληρώσει τις οικονομικές ε, υποχρεώσεις σε σχέση με τις πληρωμές που έχουν ήδη προβλεφθεί. Τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Είναι επίσης αυτονόητο κατά την άποψή μου ότι όλες οι δεσμεύσεις ε, που έχουν ληφθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 14-20 θα πρέπει επίσης να εκπληρωθούν. Αυτό είναι θέμα νομικής φύσεως. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εκπληρώσει αυτές τις και δεν καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις του, ποια δυνατότητα προσφυγής έχουμε εμείς έτσι ώστε να πιέσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει, να σεβαστεί τις υποχρεώσεις αυτές. Επίσης, ε, είναι και ένα μήνυμα που κατά την άποψή μου πρέπει να περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή την ανησυχία και των δικαιούχων στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κανονισμός αυτός ε, ε, έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε ακόμα και αν παρελπίδα ε, προχωρήσουμε σε Brexit χωρίς συμφωνία, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καλύψει τους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, πρόκειται για σημαντικά προγράμματα όπως είναι το Erasmus Plus, όπως είναι ε, προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν, όλοι αυτοί οι πολίτες δεν πρέπει να ζημιωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Έντερ ή Έντερ Γκαντιαθάμπαλ. Όχι. Hey. Ε, Εντάξει, ήσασταν τόσο σύντομη; Δεν θέλετε το λόγο τελικά. Ο κύριος Κόλμερ, ο κύριος Ντεπρέ, ούτε αυτοί έχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Σολέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είναι απίστευτο ότι συζητάμε πλέον σήμερα ένα έκτακτο σχέδιο σε σχέση με τις δεσμεύσεις ε, του προπολισμού των, Βρετα... των Βρετανών προς τον προπολισμό του 2019. Ε, εντάξει, σημαίνουν αυτά στην πολιτική διαπραγματεύση. Σας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τελικά ένα Brexit συντεταγμένο, αλλά το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα ένα τέτοιο κατεπήγον σχέδιο είναι εξαιρετικά λυπηρό. Δύο ερωτήσεις, κύριε Πίτροπε είπατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο να συνεχίσει να συνεισφέρει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε κάθε περίπτωση. Ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων, των υποχρεώσεων ε, του παρελθόντος. Μπορείτε λίγο να το διευκρινίσετε αυτό. Ποιες, ποιες ακριβώς αυτές οι υποχρεώσεις ε, στο διεθνές δίκαιο. Και δεύτερον, ποια μέτρα θα παίρνατε εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να μην σεβαστεί τις δεσμεύσεις του για τον προπολογισμό του 2019. Ευχαριστώ κυρία η κυρία Μυριάντα, συγγνώμη. Ναι, έχω πολλά να πω για το Brexit. Ε, και εγώ είμαι αισιόδοξη αλλά γενικά, αλλά τώρα εδώ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είχαμε μια συμφωνία με το Μεροσύλλο, έτσι νομίζαμε. Ε, τώρα βλέπουμε ότι αυτοί δεν την αποδέχονται τη συμφωνία αυτή και είναι αρκετά ρεαλιστικό να θεωρήσει κανείς ότι δεν πρόκειται να σεβαστούν τη συμφωνία. Και αυτό το σχέδιο, το επίγον, εξαρτάται από τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε και για αυτήν την ε, δυνατότητα, ό,τι και αν λέει το διεθνέ δίκαιο. Ξέρουμε τι μα δείχνει το παρελθόν. Ε, δεν, φτάνει, δεν φτάνουν αυτέ τι διασφαλίσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον βραχυπρόθεσμο προπολογισμό, αλλά και με τον μακροπρόθεσμο. Ακόμα και αν συμφωνήσουμε, αν συμφωνήσουμε το 2000, μέχρι το τέλο του 2019, τι θα γίνει το 2020. Όπω ξέρετε, πολλέ επιχειρήσει ε, κάνουν σχέδια τριετή, πενταετή και αυτή η αβεβαιότητα θα είναι σίγουρα επιβλαβής επιζήμια για την ε, οικονομία μας. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των ε, συμπράξεων. Ε, το, η Ιρλανδία έχει πολλές εμπορικές συμπράξεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά το 2019. Πρέπει πραγματικά να είμαστε ρεαλιστές. Είναι πιθανό τελικά οι Βρετανοί να μην συμφωνήσουν, παρότι εμεί θα θέλαμε να συμφωνήσουμε. Για λόγου λοιπόν νομική ασφάλεια θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει σε δικαίου, διότι αν δεν υπάρχει μια σαφή δέσμευση ε, σε ό,τι αφορά την ε, απόσυρση αυτή του Μένου Βασιλείου, μπαίνουμε εδώ σε ε, βάδιστα εδάφη και θα είναι εξαιρετικά περίπλοκα τα πράγματα. Θα πρέπει να συζητήσουμε δηλαδή τι θα συμβεί εφόσον οι Βρετανοί δεν συμφωνήσουν. Και θέλω να απάντηση για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Merci. Ο κύριος Αρνότ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή ε, σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη στον Μενοβασίλειο. Ε, αν δείτε το δημοψήφισμα του 2016, τότε την εκστρατεία την ε, προεκλογική. Κάποιοι έλεγαν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση που το Ευρωπαϊκό Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάνουν σε συμφωνία. Ε, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίω θα ήταν υπέρ μια συμφωνία παρόλα αυτά. Αυτό όμω που διαπιστώνουμε τώρα είναι ότι λόγω τη κατάσταση με τι διαπραγματεύσει και βεβαίω θα αποκλίνουν οι απόψει μα, φαντάζομαι, για το πώ φτάσαμε εδώ, αλλά εν πάση λόγω τη κατάσταση που είναι διαπραγματεύσει τώρα αυτή τη στιγμή, έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι όχι μόνο δέχονται την πιθανότητα της μη συμφωνία, αλλά που θέλουν να μην υπάρξει καμία συμφωνία. Ε, και είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει το 30% στι δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ε, ε, το Κοινοβούλιο με μικρή πλειοψηφία είπε ότι ε, δεν είναι κατά του... Είναι κατά, δεν δέχεται να μην υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Αυτός ο προτινόμενος κανονισμός, πάντως, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ειδωθεί όσο ότι θα πληρώσουν ε, 17 δις ε, στο κοινωνικό προπολογισμό ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία. Ε, για το Brexit. Και αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ε, θα το υποδεχθούν πολύ άσχημα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και ως κάτι ουτοπικό στην πραγματικότητα. Το να συμφωνεί στον Ηνωμένο Βασίλειο σε κάτι τέτοιο δηλαδή. Και κάτι άλλο τώρα. Σε σχέση με τον κανονισμό, ένας ξεχωριστός κανονισμός από ό,τι κατάλαβα, που υπάρχει. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει, συμφωνήσει μάλλον για το, τις προϋποθέσεις του Εράσμους, αλλά όχι γι' αυτό τον κανονισμό. Θα είναι διαφορετικά νομοθετήματα ή ισχύει το ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τίποτα αν δεν υπάρχει συμφωνία για τα πάντα. Σας ευχαριστώ. Όσοι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, τώρα θα τον έχουν. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε την διαφορά ανάμεσα στην συμφωνία από δημοσιονομική πλευρά την ε, συμφωνία που αφορά το 21, 22 και 23. Η συμφωνία που προετοιμάστηκε δείχνει ότι το ε, Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να παραμείνει στον προϋπολογισμό, αλλά σε όλα τα προγράμματα μέχρι το 2020. Το ερώτημα που προκύπτει δεν αφορά μόνο τον προϋπολογισμό, αλλά και τη λειτουργία των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ηνωμένου Βασιλείου. Από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε μην ανησυχείτε, θα υπάρξει κάποια λύση. Δηλαδή, στην ουσία δεν συζητούμε την σχέση με, εντός της Ευρωπαϊκής Μιλάμε για μια πρόσκαιρη λύση μεταξύ δύο απολύτως ανεξαρτήτων οντοτήτων. Από τη μία πλευρά έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και από την άλλη πλευρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των δύο ε, υπάρχει μια ε, πρόσκαιρη λύση. Όσον αφορά τώρα την πρόσκαιρη λύση, εάν ε, μιλάμε για την Βρετανική συνεισφορά στον ε, ενωσιακό προϋπολογισμό του 19 και θυμάμαι εδώ τις πληροφορίες που είχαμε ότι την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους θα η υπογραφή, η συμφωνία ε, και το συμβόλαιο για δύο μέρες, γιατί μετά από δύο μέρες θα πρέπει να φύγουν, θα πρέπει όλα να λυθούν, ε, να υπολογιστεί μισθός, ε, φόροι κλπ. για δύο μέρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει τον Μάρτιο, αλλά ερώτηση, τα κράτη-μέλη... Έχουμε την επιστροφή και τι θα γίνει, ε, θα συμφωνήσουν ε, τα κράτη-μέλη, ε, διότι... Άλλο θα πληρώσει 11 συγκεκριμένα χωρίς επιστροφή και 17 με επιστροφή. Δεύτερον, συζητούμε για πληρωμές ή... ή μιλάμε για υποχρεώσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλές ε, ε, ε, επενδύσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, προγράμματα που τρέχουν και ε, φυσικά εάν ε, μιλάμε για πληρωμές είμαστε, είναι σαφές πρέπει να ε, προχωρήσουν. Οκ, αλλά συμφωνώ τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις για το 2019. Έχουμε συμφωνήσει, εάν συμφωνήσουμε για τις δεσμεύσεις το, του, 2019, τις υποχρεώσεις του 2019, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε συμφωνία για την εκτέλεση που θα γίνει το 2020 και επομένως τότε θα πρέπει να πληρώσουν όλοι διαφορετική συνεισφορά. Και δεν νομίζω ότι η Γαλλία πούμε, θα συμφωνήσει να πληρώσει 1,5 δις. Τι γίνεται λοιπόν με τις δεσμεύσεις ε, ε, υποχρεώσεων. Πιστώσεις υποχρεώσεων. Ε, γιατί θα ολοκληρωθούν, εάν συμφωνήσουμε από αυτόν, θα ολοκληρωθούν το 2020. Και αν δεν υπάρχει συμφωνία θα έχουμε πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει κατά κάποιο τρόπο και με τον έρασμο θα προχωρήσουμε σε τελείως νέα σύμβαση στην ουσία. Γιατί κάποια στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία και ξαναρχίζει με νέο τρόπο. Βεβαίως είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά εν συνόψη τι γίνεται με τις επιστροφές και τι γίνεται με τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Um, Mr. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλη αυτή η ιδέα του no deal Brexit, Brexit χωρίς συμφωνία, είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Πιστεύω ότι είναι μια μπλόφα στην ουσία. Είναι μια μπλόφα στην ουσία η οποία στόχο έχει να διασφαλίσει ότι ε, θα σκεφτούν ε, ε, το μη χειρον βέλτιστον οι κάτοικοι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα, σε σχέση με την καλύτερη δυνατή συμφωνία που είπε, που ανέφερε ο κύριος Επίτροπος, είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει στη διαπραγμάτευση το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αν είχε γίνει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση θα μπορούσαμε να είχαμε μια τελείως διαφορετική διαφορετική κατάσταση. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ε, ε, καμία ε, περίπτωση αναχώρησης τέτοιου είδους δεν θα, δεν, θα είχε κατά νου η Βρετανία ήδη από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι έτοιμο για μία αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι ήδη μέχρι σήμερα, μέχρι χτες έπαιρναν κονδύλια από συγκεκριμένα προγράμματα και που έχουν τεράστια ασάφεια ε, γιατί δεν έχουν την δυνατότητα συνέχισης των πιστώσεων και δεν έχουν δυνατότητα αυτόνομης ε, ε, κίνησης και επίσης το θέμα δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασιλείο γιατί είναι πολύ μεγάλη η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις, στα, στα θεσμικά όργανα, στους θεσμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ οπωσδήποτε θα πρέπει ε, ε, να ε, ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα το οποίο ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε προκύψει γιατί εάν οι πολιτικοί ενδιαφέροντο για σοβαρά πράγματα και όχι μονάχα για τα τυπικά γιατί βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες, στους ερευνητές, πώς θα συνεχίσουν τα ερευνητικά κέντρα και οι επιστήμονες στη το, η Πρωθυπουργό ε, ε, στις δηλώσεις που έκανε ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Ε, ε μερικοί την παίρνουν κατά γράμμα, εγώ όχι τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις οπωσδήποτε. Ξεκαθάρισε ο ε, κ. Επίτροπος προηγουμένως ότι υπάρχουν υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν ε, βάσει υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές ε, δίκαιο. Πρέπει να πούμε τώρα, εάν όλα αυτά τα στοιχεία, η ερμηνεία του νόμου και η ερμηνεία που δίνει και η Πρωθυπουργό δεν θα πρέπει να οδηγήσει οπωσδήποτε στην υπογραφή αυτή τη συμφωνία, γιατί διαφορετικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποφέρει πάρα πολύ. Η φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου θα υποφέρει πάρα πολύ. Ε, και εδώ παίζεται η αξιοπιστία και ε, η φήμη και η πολιτική σταθερότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και επομένως πιστεύω ότι μονόδρομος είναι η προσυπογραφή, η συμφωνία. Ε, και όταν ε, ε, θα προχωρήσει η Κομισιόν και τη συγχαίρω γι' αυτό όταν θα προχωρήσει αυτό το Plan A γιατί πραγματικά δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τέλη Μαρτίου να προχωρήσουμε σε Plan B. Ευχαριστώ κυρία Αλμέιερ έχει το λόγο. Κυρία μετά τα όσα είπε ο Γιάνν Όλμπριχτ θα είμαι σύντομη. Το βασικό μου ερώτημα έχει ως εξής τι θα κάνουμε εάν έφνης η Μεγάλη Βρετανία αποφασίσει στις 29 Τρίτου να σταματήσει τις πληρωμές και να θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται από τίποτα. Έχω απόλυτη κατανόηση για τις θεωρίες που εξήγησε μόλις ο Βρετανός συνάδελφος, αλλά για να είμαι ειλικρινής, μετά από τις συζητήσεις που παρακολούθησα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τις οποίες ε, παρακολούθησα με κάποια έκπληξη, Βεβαίω έχουν κάπω χιουμοριστικό χαρακτήρα ορισμένε φορέ, αλλά εάν δεν γνωρίζει κανεί ε, τι κοινοβουλευτικέ αυτέ συζητήσει, το βρίσκει και λίγο αστείε. αλλά νομίζω ότι η Βουλή των Κοινοτήτων συμφωνεί στο ότι διαφωνεί. Δεν είναι υπέρ ούτε του σκληρού Brexit, ούτε υπέρ του μαλακού Brexit, ούτε υπέρ νέων διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, εν τέλει, συμφωνούν ότι θέλουν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουν όσο γίνεται λιγότερα. Αυτό διαπιστώνω εγώ. Και εάν καταλήξει κανεί πράγματι σε αυτό το συμπέρασμα, θα ήθελα να μάθω εγώ ποια είναι τα σχέδια των χώρων μελών για την περίπτωση ότι μέχρι το τέλο του 2019 θα γίνει απολύτω τίποτα και δεν θα καταβληθούν καθόλου χρήματα από το Ηνωμένο ή πολύ λίγα ομολογώ ότι η φαντασία μου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Θα ήθελα να με μιλήσετε λίγο περισσότερο στα ενδεχόμενα σενάρια τα οποία έχετε. Merci. Monsieur Rubig. Κύριε Ρούμπικ, ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Μόνο την 1η Απριλίου θα γνωρίζουμε, αυτό είναι το γεγονός, τι θα γίνει ακριβώς. Ή έστω και λίγο αργότερα, όπως λέει κάποιος που δεν έχει μικρόφωνο. Σύντομα θα δούμε όμως και τις συνέπειες, τις επιπτώσεις. Το ερώτημα είναι θα υπάρξει άλλο δημοψήφισμα. Όχι, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει η συμφωνία της αποχώρησης. Αν απορριφθεί, τελος πάντων, αν υπάρξει νέο δημοψήφισμα, εν πάση περιπτώσει, θα παραμείνει τότε ε, χώρα μέλος η Μεγάλη Βρετανία και αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα. Τώρα, κάνει η κυβέρνηση, η Βρετανική κυβέρνηση μια συμφωνία και μετά το κοινοβούλιο δεν την δέχεται για δύο λόγους. Αφενός όσοι θέλουν το σκληρό Brexit, αυτό σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία στην περίπτωση αυτή, δηλαδή μη συμφωνίας, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στο καθεστώς του Ουσβεκιστάν. Δηλαδή, λέγαμε πριν ότι μπορεί να είναι Αυστραλία ή Νέα Ζηλανδία. Όχι, αυτές οι χώρες έχουν διμερεί συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα Γι' αυτό το Ουσμπεκιστάν είναι το παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Το ερώτημα είναι μετά τι κάνουμε με τη Βόρεια Ιρλανδία. Νομίζω ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα γίνει και αυτή πια τρίτη χώρα. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τις πληρωμές στην Βόρεια Ιρλανδία ως τρίτη χώρα. Γιατί θεωρώ ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα χρειαστεί απολύτως υποστήριξη. Για μένα είναι σαφές επίσης ότι εν τω μεταξύ η Ελβετία έχει διαπραγματευτεί με την ε, Μεγάλη Βρετανία και στην βάση και των δύο σεναριών, δηλαδή και στην βάση της χαούδους αποχώρησης, αλλά και στην βάση της διδεταγμένης με συμφωνία. Η Ελβετία λοιπόν έχει ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει αυτό συνέπειες για εμάς. Και το ερώτημα επίσης είναι, επειδή είμαι αρμόδιος για τους οχτώ οργανισμούς που θίγονται η αποχώρηση των ευρωβουλευτών σημαίνει ότι στην περίπτωση που παραμένουν Ευρω... Ε, Βρετανοί ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Τι γίνεται, ε, για παράδειγμα, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποιοι θα αποχωρήσουν την 1η Απριλίου. Ποια μέλη ποιων θεσμών. Και με τις ε, σημαίες μεσίστιες την 1η Απριλίου θα αποχαιρετήσουμε ποιους Βρετανούς φίλους. Είναι εξάλλου σαφές ότι η αποχώρηση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά αναλογία όπως και οι φάσεις ένταξης. Ε, δηλαδή, για την ένταξη έχουμε μία πορεία σε φάσεις. Νομίζω για την αποχώρηση μπορεί να γίνει αναλογικά το ίδιο. Και από την άλλη μεριά, ο προϋπολογισμός του 2019 έγινε αντικείμενο διαπράγματευση ήδη με τη Βρετανική κυβέρνηση. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο η Βρετανική κυβέρνηση ε, δεν είναι διατεθειμένη να σεβαστεί τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Ήταν σαφέ όταν ενέκρινε τον προπολογισμό αυτό ότι εκινείται η διαπραγμάτευση για την αποχώρηση. Ήταν καθαρό επίση ότι ενδέχεται να υπάρξει hard Brexit. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπολογισμό αυτό θα πρέπει να μπορεί να εκτελεστεί και ότι επομένω πληρωμέ ε, πιστώσει μάλλον υποχρεώσεων και πληρωμών θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ και να εκτελεστεί ο προπολογισμό. Είναι και ζήτημα εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να κάθεται κανεί και να συζητεί γνωρίζοντα ότι είναι δυνατό να γίνει και hard Brexit και ξαφνικά να αποφασίσει ότι σταματά τις ε, πληρωμές είτε υποχρεώσεων είτε τις πιστώσει, μάλλον. Αυτό δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να δεχθούμε δηλαδή η κατάσταση του Ουσμπεκιστάν. Ευχαριστώ, κύριε Βάλλη. Πολύ σύντομα κι εγώ. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις εντάχει. σε σχέση με αυτό που είπαν συνάδελφοι, ναι, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια και σχεδιασμοί για περίπτωση μη συμφωνίας. Ε, ε, προσθέτω δε ότι εγώ ήμουν ε, εισηγητής για τον προϋπολογισμό 2019 και αν δεν υπάρχει συμφωνία θα το πάρω πολύ προσωπικά. Θα είναι προσωπική προσβολή για μένα και θα θύμωνα πολύ. Αλλά πέρα από το θυμό και αν δεν υπάρξει συμφωνία, πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι ε, αυτό αυτό το ε, πολύ μικρό χρονοδιάγραμμα ε, μας δίνει τη δυνατότητα ε, να υπάρξει έγκριση ε, σε εθνικό επίπεδο από τα εθνικά κοινοβούλια. το, έχουμε το, τη συνάντηση των Υπουργών Γενικών Υποθέσεων τον Μάρτιο, αλλά έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν βέβαια και το δίκαιο σε περίπτωση μη συμφωνίας. Επίσης, τι ε, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα πρέπει να είναι το 100 ε, εκατομμυρίων ε, και πότε θα πρέπει να υποβληθεί. Ευχαριστώ κυρία Τωμά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν σας άκουσα κιόλας οπότε ενδεχομένως να πω και κάποιες βλακίες ε, εν πάση περιπτώσει για το θέμα αυτό του Brexit. Εγώ συνήθως ε, συνηθίζω πάντα να σκέφτομαι το χειρότερο ε, και μετά βεβαίως είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. και πρέπει να σκεφτούμε και τα χειρότερα στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον σε ό,τι δύο θέματα που αφορούν και την περιοχή από την οποία προέρχομαι, τα λιμάνια και η αλία. Στον τομέα της αλίας, εάν δεν υπάρχει συμφωνία, σε πολλές περιοχές, και τουλάχιστον 6-7 χώρες της Ένωσης, κάποια πλοία ε, τα οποία αλλιεύουν στα Βρετανικά ύδατα δεν θα μπορούν πλέον να το πράξουν. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν και να ψαρέψουν στα ευρωπαϊκά ύδατα, μιας και υπάρχει ήδη σημαντική πίεση στους πόρους εκεί, την οποία δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να αυξήσουμε, δηλαδή την αληφτική δραστηριότητα. Θα υπάρξει βεβαίως μια τροποποίηση του Ταμείου, γύρω στο, στο, του Ταμείου στην Επιτροπή Αλίας, αλλά πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά το ζήτημα αυτό, διότι εάν κάποιοι δεν μπορούν να ζήσουν από την εργασία τους, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ε, να τους πλαισιώσουμε ενδεχομένως ε, ε, σε ένα παναπασαντολισμό της εργασίας τους κτλ. Ε, λέω απλώς ότι πρέπει να, γίνει, να υπόψη το θέμα της αλίας και κάτι άλλο τώρα για τα λιμάνια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία, έχουμε να κάνουμε μια τρίτη χώρα. με τελωνία, εκτελονισμούς, ε, ιατρικός έλεγχος για τα ζωικά προϊόντα και για τα τρόφιμα ενδεχομένως. Ε, οπότε αυτό αλλάζει τα πάντα για τα λιμάνια της Βρετάνης, ας πούμε, της Βόρειας Γαλλίας, αλλά φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για το Βέλγιο, ε, για τις κάτω χώρες, Σουηδία, Δανία. είναι σαφές ότι για αυτά τα λιμάνια θα πρέπει οι υποδομές να προσαρμοστούν. Διότι συνήθως όταν φτάνουν τα φέρι ε, στη χώρα μας βγαίνουν οι επιβάτες στα φορτικά χωρίς έλεγχο, έτσι, από την Αγγλία. Από που έχουμε να κάνουμε μια τρίτη χώρα όμως, ε, αλλάζουν τα πράγματα. Ήθελα απλώς να αναφέρω αυτά τα δύο σημεία τα οποία είναι σημαντικά. Ε, το ίδιο ισχύει για τα αεροδρόμια. Τώρα εντάξει, να μην τα πω όλα. Υπάρχει ένα αεροδρόμιο κοντά στο σπίτι μου, μικρό, που ουσιαστικά εξυπηρετεί πτήσει μόνο προ και από την Αγγλία, τον Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήδη αυτά τα θέματα τα έχετε σκεφτεί, αν τα αναφέρατε. Φαντάζομαι τα κράτη-μέλη τα ίδια ε, τα έχουν σκεφτεί, αλλά Εάν κάνουμε αυτό τον κατάλογο με όλα αυτά τα μέτρα, προποθέτουν ένα δημοσιονομικό κόστο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Έχω και δικό δύο ερωτήματα όμω. Επιπλέον, πριν από δύο εβδομάδε στο Στρασβούργο, ο κ. Σέλμαιερ ήρθε στου επικεφαλεί των επιτροπών και σε κάποιου εισηγητέ και αναφέρθηκε στα επίγοντα μέτρα που θα παρθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση μη συμφωνίας. Και εμείς είχαμε καταλάβει ότι από την οικονομική πλευρά δεν θα υπάρξει κάποιος αντίκτυπος. Τις επόμενες μέρες, διαβάζοντας το πολίτικο, μάθαμε ότι η Κομισιόν θα περιορίσει ε, τις ε, δεσμεύσεις και τις πληρωμές ε, για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση σε περίπτωση μη συμφωνίας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι από αυτού. Και κάτι άλλο τώρα. Σχετίζεται και με τα σχόλια όλων. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε πολιτικούς ηθήνοντες υποψήφιους ε, που επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προεκλογικά, λένε ότι θα φύγουν από την Ευρωζώνη και μόλις εκλεγούν, ε, βολευόμαστε με τις διατάξεις της Ένωσης και με την Ευρωζώνη. Είδαμε πριν από τέσσερα χρόνια ένα πρωθυπουργό που για έξι μήνες ε, δεν συμφωνούσε με τη συμφωνία των πιστωτών, οργάνωσε δημοψήφισμα, ο λαός ψήφισε κατά τη συμφωνίας και ο Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα υπέγραψε τη συμφωνία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση, μια ανθεκτικότητα οικονομική, νομισματική και που αρχίζει να υπάρχει και σε κοινωνικό επίπεδο το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να, να νιώσει αυτή την, βρετανική, την ευρωπαϊκή συγγνώμη ανθεκτικότητα. Ε, ενδέχεται λοιπόν εφόσον έχουμε έτσι δραματικές επιπτώσεις περί του σημείς συμφωνίας να, να ακουστούν κάποιες φωνές από την άλλη πλευρά της μάχης για μια παράταση. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ένωσης. Και μπορεί να έχουμε και υποψήφιους ε, για τις ευρωεκλογέ. Η Κομισιόν τι πιστεύει από αυτού. Μια παράταση δηλαδή έως ε, την οργάνωση κάποιου άλλου δημοψηφίσματος στο Μένο Βασίλειο ε, για την οριστική έξοδο ή τη διατήρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Επίτροπος Έτιγκερ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας που είναι πραγματικά θεμελιωμένες σε γνώση και που αναφέρονται εν μέρη στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019, αλλά υπερβαίνουν και όλα στα όρια αυτά. Για την απάντηση των ερωτήσεων που δεν άπτονται του προϋπολογισμού δεν είμαι πραγματικά αρμόδιος. Παρ' όλα αυτά θα τοποθετηθώ εν συντομία. Εάν η Βρετανική πλευρά ζητήσει παράταση, δηλαδή αναβολή τη αποχωρησεω κατα κατά δύο-τρει μήνε και υπάρξουν λόγοι, υπάρχουν πραγματικοί λόγοι, βλέπω πραγματικά τη δυνατότητα οι χώρε μέλη, να, οι υπόλοιπε χώρε μέλη, δηλαδή να αποδεχτούν την, το αίτημα αυτό ομόφωνα. Όμως θα πρέπει να υπάρχει η πραγματική ουσιαστική πιθανότητα να υπάρχει πρόοδος και να υπάρξει εν τέλει μια συμφωνία αποχωρήσεως. Τώρα, μακρότερη παράταση σημαίνει ότι συγκρούνται πλέον, πλέον με τις ευρωεκλογέ. Η χώρα μέλος θα πρέπει να σεβαστεί και να εγγυάται το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Αν τώρα ενδεχομένως υπάρξει άλλη λύση, δηλαδή απόσπαση ε, βουλευτών όπως έγινε και στην περίπτωση της Γερμανικής ε, Επανένωσης. Όμως τότε ήρθαν για τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περίοδου ένας αριθμός 18 εκατομμυρίων νέων Ευρωπαίων πολιτών. Και οι βουλευτές που αποσπάστηκαν τότε ήρθαν, συμμετέσχουν μετά στις ευρωεκλογέ. Όμως η Βρετανία εξακολουθεί να είναι χώρα μέλος. Δεν υπάρχει λόγο λοιπόν να μην συμμετάσχει στι ευρωεκλογέ εάν υπάρξει παράταση κατά δύο ή τρει μήνε. Τώρα, το ζήτημα τη ε, της είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι μιλούμε για ψαράδε από Γαλλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Δανία. Ψαρεύουν σε χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου εφόσον πρόκειται για ενιαία αγορά για να μπορέσουν λοιπόν να ασκήσουν την επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτή η δυνατότητα εκπίπτει άμεσα εάν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό είπε πάντοτε και ο Μισελ Μπαρνιέ ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα αλίας, αυτό θα είναι προσφορά των Βρετανών προς εμάς, που θα μπει σε ένα πακέτο και θα χρειαστεί μια αντιπαροχή δική μας προς τους Βρετανούς. Άρα θα πρέπει να μπει στα πλαίσια μιας συμφωνίας Δούνε και Λαβίν. Το ίδιο τώρα. Αερολιμένες και η αναγκαία έλεγχη. Εκεί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερεπιβάρυνση των διοικήσεων και να υπάρξει κίνδυνος χαόδου εξελίξεως. Ο πρόεδρος διακόπτη. Ναι, ε, βεβαίως ε, οι αλλιευτικές ε, περιοχές είναι βρετανικές. Από την άλλη μεριά όμως οι ε, Βρετανοί αλληλείς ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά ε, γιατί πουλάνε την, ε, το αλλήλευμά τους στην ευρωπαϊκή αγορά άρα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στους αλληλείς και τους καταναλωτές. Αν καταλήξουμε σε αποχώρηση χωρίς συμφωνία και οι αλληλείς πλήττονται στην επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε από την κοινή γεωργική πολιτική να διαθέσουμε έκτακτα κονδύλια για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να αποφύγουν την πτώχευση. Να τους υποστηρίξουμε δηλαδή οικονομικά ώστε να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τα μειονεκτήματα που θα προκύψουν από την αποχώρηση. Θα γίνει τώρα αν δεν υπάρχει συμφωνία. Εγώ δεν θέλω να οικοτολογήσω. Είναι σαφές πάντως ότι εάν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο αυτό, θα ήταν μεγάλο λάθος μας. Η πιθανότητα να υπάρξει αποχώρηση χωρίς συμφωνία δεν είναι μηδενική. Εγώ την υπολογίζω στο 30 με 60% και των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε το contingency plan για τον κοινωνικό τομέα, για τον συν και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αυτά τα βάζουμε σε, ως μια πρόταση στους Βρετανούς και περιλαμβάνουμε όλους τους οικονομικούς τομείς, όλες τις εισαγωγές-εξαγωγές, όλες τις παροχές υπηρεσιών. Τα αναλύσαμε όλα αυτά και τα έχουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι τον Μάρτιο, αλλά ήδη από σήμερα. Μέσω των οργανώσεων, της οικονομίας μέσω των επιμελητηρίων, μέσω των ε, μέσων ενημέρωσης θα παράσχουμε πλήρη ενημέρωση σε όλους όσοι συμμετέχουν στην οικονομία των 27 χωρών μελών και θα δώσουμε συγκεκριμένες συμβουλές για το τι να πράξουν. Αυτές βρίσκονται στην φάση της προπαρασκευής και μάλιστα είναι πολύ προχωρημένη η προπαρασκευή αυτή. Οι δε υπηρεσίες μας κάνουν συγκεκριμένες αναλύσεις για τη μείωση των ζημιών ανά τομέα. Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει μερικώς τους κανονισμού μας, γιατί η δικαίωμά του είναι, το Συμβούλιο είναι εν προκειμένου ο νομοθέτης και εσείς ως Κοινοβούλιο καλείστε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε τον κανονισμό. Εάν δηλαδή το, το Συμβούλιο εγκρίνει μόνο το τμήμα του έρασμο συν. Καλύτερα από το τίποτα. Εάν τώρα οι Βρετανοί από τα πακέτα για την έρευνα, γεωργία, κοινωνικά, έρασμο, θελήσουν να πάρουν μόνο ένα τμήμα, θα πρέπει εμείς τότε να κρίνουμε αν το θεωρούμε αυτό αποδεκτό ή όχι. Θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε ποια τμήματα δέχονται οι Βρετανοί φίλοι μας και ποια όχι. Το ίδιο για τις επιστροφές. Το Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τις επιστροφές ή εάν εκπίπτουν οι επιστροφές για το Αμένο Βασίλειο άμα τη αποχωρήσει. Η, η ε, πρότασή μας αναφέρεται και στις πιστώσεις υποχρεώσεων και στις πληρωμές. Πολλές από τις πληρωμές του 2019 για το έρασμο συν δίνουμε χρήματα στους νέους μήνα, κάθε μήνα για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Πρόκειται δηλαδή για υποχρεώσεις και πληρωμές που είναι σχεδόν ταυτόσιμες χρονικά. Για μεγαλύτερα έργα οι πληρωμές συνεχίζονται και για μεγάλο διάστημα μετά από την εξάρτηση των υποχρεώσεων. Είναι ορθό, και το επαναλαμβάνω, ότι από τη σκοπιά του καθαρού συνεισφορέα η προσφορά μας δείχνει ότι οι Βρετανοί μας φίλοι θα πληρώσουν κάτι παραπάνω για το 2019 από ότι θα λάβουν επιστροφές από τον προϋπολογισμό μας για τα προγράμματα. Όμως, αυτό σημαίνει ότι τα Βρετανικά ερευνητικά κέντρα και οι Ινστιτούτα, οι γεωργοί τους, οι νέες και νέοι τους, θα αποφύγουν το χάος. Αυτό θα πρέπει να το κρίνει η πολιτική ηγεσία στο Λονδίνο. Τι είναι πιο σημαντικό για αυτού. Σίγουρα θα παίξει και ένα ρόλο ποια θα είναι η ατμόσφαιρα των σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών. Εάν είναι δηλητηριώδη, τότε οι σκληροπυρηνικοί του Λονδίνου θα απορρίψουν την πρότασή μα. Εάν υπάρχει μια συναντριφική ατμόσφαιρα παρά τι διαφορέ απόψεων, θα την αποδεχτούν. Όμω η πρόσφορα που κάνουμε εμεί και η πρόταση που απευθύνουμε προ Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να μην είναι αποδεκτή, αυτό ήταν λάθο. Κατά βάση, πρόκειται για μια μικρή συμφωνία αποχώρηση. Περιορίζεται στον προπολογισμό, περιορίζεται στα προγράμματα και περιορίζεται στο 2019. Πρόκειται για ένα μικρό λιθαράκι, το οποίο εντάσσεται σε. Θα, θα εντασσόταν κανονικά σε μια ευρύτερη συμφωνία αποχωρήσεως. Αυτή είναι η προσφορά μας ένα μίνι, μια μίνι συμφωνία αποχώρησης δηλαδή στην πραγματικότητα. Το ερώτημα τώρα, εάν δεν πληρώσουν οι Βρετανοί, παρόλο που έχει εγκριθεί ο προπολογισμό του 2019 και παρόλο που το δημοσιονομικό πλαίσιο πηγαίνει μέχρι το 2021, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι τότε παραμένουν μονάχα οι διεθνεί δικαιοδοσίε, τα διεθνή δικαστήρια. Δηλαδή, όπου θα πρέπει να προσφύγουμε για να εξασφαλίσουμε τις πληρωμές μέχρι ε, το τέλος του 2020. Αλλιώς βέβαια θα είναι η τελική κρίση, ας το πούμε έτσι, η ημέρα της κρίσεως. Τώρα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών νομίζω θα ψηφίσει 18 Τρίτου και θα δώσει σύμφωνη γνώμη ή απόρριψη 3 με 4 Απριλίου. Και το Συμβούλιο Πριν από αυτό θα πρέπει να έχει εξετάσει σε ομάδες εργασίας το, ε, την πρότασή μας το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εγκρίνει 18 Απριλίου, μετά από δηλαδή το Κοινοβούλιο. Οπότε θα έχουμε μία προσφορά η οποία θα είναι νομικά εγκεκριμένη προσφορά 9 μέρες πριν από την τελική ημερομηνία αποχώρησης. Και οι Βρετανοί έχουν τότε τη δυνατότητα μέχρι τις 30 Απριλίου να αναλάβουν τη σχετική υποχρέωση να δεχθούν τους οικονομικούς ελέγχους κλπ. Και νομίζω για να γίνει η καταβολή της πρώτης δόσης της συνεισφοράς τους είναι νομίζω η 8η Απριλίου. Απάντησα στα πιο θεμελιώδη ερωτήματα. Κατά τα άλλα, οι ερωτήσεις που υποβάλλονται και στην ομάδα εργασίας άρθρου 50 και οι γραπτές σας ερωτήσεις, μάλλον οι ερωτήσεις σας, τις οποίες θα απαντήσουμε γραπτός, θα χρειαστούν τρεις εργάσιμες ημέρες. Θα τις λάβετε λοιπόν αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπη για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ε, μας διαφωτίσατε με τις ε, ε τοποθετήσεις σας ε, για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν θα που θα αποχωρήσει το ΕΒ Βασίλειο χωρί συμφωνία στι 29 Μαρτίου. Ε, αυτό το σχέδιο κανονισμού ε, ισορροπεί μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων που ε, θα πλήξουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΒ εφόσον ε, το ΕΒ Βασίλειο ε, δεν σεβαστεί τις δεσμεύσεις του ε, αυτό είναι κάτι βεβαίω ε, που θα πλήξει τον Ηνωμένο Βασίλειο και την φήμη του ε, παγκοσμίω και από εκεί πέρα τα αντίπεινα θα ήταν να σταματήσουμε οποιαδήποτε πληρωμή ε, ως Ευρωπαίοι προς βρετανικά συμφέροντα, βρετανικές επιχείρησει Ε, κοινή λογική λέει ότι θέλουμε να αποφευχθεί αυτό ο κατακλυσμό. Ε, ε, το καλύτερο θα ήταν μάλιστα να υπάρξει αναβολή, αυτό, αυτό πιστεύω. Θα δούμε τώρα το Μάιο τελικά εάν οι Βρετανοί εκλογής ε, οι Βρετανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να εκλέξουν ε, βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, είμαστε σε συνεχή επαφή. Euh, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον αρνητικό αντίκτυπο στην εκτέλεση του προπολογισμού 2019, ε, ο Γενικός Συγητής και οι συγητές ε, των άλλων τμήματων θα επαγρυπνούν, όμως μπορούμε ήδη να συζητήσουμε και το 2020, διότι και αυτό είναι ένα σημείο ανησυχίας. Και για να μας φωτίσει για το τι θα συμβεί το 2020 και τον προπολογισμό θα δώσω το λόγο στον, στην Μόνικα Ολμέγερ ευχαρίστως γενική συγκίτρια, της οποίας η πανεκλογή στο Κοινοβούλιο είναι δεδομένη για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι γενική συγκίτρια και μετά την 1η Ιουλίου Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, πράγματι οι προοπτικέ ε, είναι καλέ να επανεκλεγώ. Τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι ψηφοφόροι. Αυτό ισχύει για όλες και όλους μας. Παρ' όλα αυτά, σε εγγύψουμε στα σοβαρά και με προσοχή στον προπολογισμό του 2020 και για τον λόγο αυτό έχω κάνει και πρόταση για τις guidelines Ήδη εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη που δεν έχω μπορέσει να τα ε, ε, χειριστώ όλα με απόλυτη ακρίβεια. Βεβαίως θα συνεχίσουμε με τροπολογίες συμπλήρωσης και τροποποίησης γιατί βέβαια το χρονικό διάστημα που μας διατίθεται δεν αρκεί για να ασχοληθούμε και με θέματα ε, αναπτυξιακής βοήθειας κλπ. Όπως είπε ο κύριος, μάλλον όπως γνωρίζει ο κύριο Βιώτη, είμαστε υποχρεωμένες να περιοριστούμε σε αυτό που είναι δυνατόν σε μια πρώτη φάση. Και μετά σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και θα συμπληρώσουμε το σχέδιο προπολογισμού έτσι ώστε τελικώ να περιλάβει όλα όσα επιθυμούμε. Στις guidelines τώρα για φέτος προσανατολίστηκα και στα όσα άρχισε ήδη από πέρυσι ο κύριος Βιώτη, διότι τα κέντρα βάρους που ε, ε, αποφασίζουμε δεν αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο, αλλά εντάσσονται και μέσα στη λογική της συνέχειας του προϋπολογισμού και ιδίως στοχεύουμε ιδίως σε θέματα ορίζοντα 2020 καινοτομία και έρευνα για τις μελλοντικέ εξελίξεις όπου περιλαμβάνεται και το σημαντικό ερώτημα το οποίο συζητήσαμε και στην τελευταία δημοσιονομική συζήτηση σε ό,τι αφορά προγράμματα τα οποία υποχρηματοδοτούνται, από την άλλη μεριά έχουν μεγάλη αποδοχή στις χώρες μέρη και συμβάλλουν σημαντικά στις οικονομίες των χωρών, όπως το κόσμε ιδίω για χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Επίσης θέματα ασφάλειας και ειρήνης, ζητήματα αλληλεγγύης και αμοιβαία κατανόησης. Εκεί τονίζω και πάλι τον έρασμο, όπου είχαμε ε, τόσο έντονα προωθήσει την τελευταία φορά και το ζήτημα του ΓΕΙ, το οποίο μας απασχολεί σε και πέρσι τόσο πολύ και που βλέπω και φέτος πώς εξελίσσονται και πώς τροποποιούνται τα προγράμματα. Εξάλλου, προβλήματα περιβάλλοντος, αλλαγής κλίματος κλπ. Τα περιέλαβα σε μία σύντομη φράση. Σας ανακοινώνω όμως από τούδε ότι, αν συμφωνήσετε και εσείς, θα κάνουμε ευρύτερες και προσεκτικότερες διατυπώσεις, γιατί είναι από τους βασικότερους τομείς, γιατί μιλώ για θέματα μεταναστευτικού και της μοίρας των ανθρώπων οι οποίοι ξεκινούν μακρές πορείες και θέλουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την μοίρα αυτή με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Σας ευχαριστώ ήδη για τις προτάσεις που μου έχετε εν μέρει ήδη υποβάλει. Αναμένω με ενδιαφέρον την συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις και υποδείξεις που μου έχετε υποβάλει αλλά και που θα μου υποβάλλετε και εύχομαι και ελπίζω όλες και όλοι μαζί να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή θέση, διότι η συζήτηση που μόλις διεξαγάγαμε τώρα πριν από λίγο δείχνει νομίζω καθαρά τι μας περιμένει ο προπολογισμό του 2020 θα είναι και ο μεταβατικό προπολογισμό ε, προ την κατεύθυνση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Την προηγούμενη φορά οι χώρε μέλη προσπάθησαν να κρατήσουν όσο γίνεται πιο χαμηλά τα κονδύλια του μεταβατικού προπολογισμού. Και θα θυμάται ο πρόεδρο, και βεβαίω ασφαλώς το γνωρίζει και ο Αλάν Λαμασούρ όπω και ο κύριος Φερνάντε, ότι τότε είχαμε αγωνιστεί και κατά των χωρών μελών οι οποίες δεν ήθελαν να καταβάλουν όλες τις πληρωμές. Και στο δεύτερο τρίτο γύρο όταν είχε εγκριθεί το ΠΔΠ είχαμε δηλώσει με αγανάκτηση ότι δεν προωθούν τις πληρωμές οι χώρες μέλη προκαλώντας έτσι μια σιωπηρή υπερχρέωση που δεν επιτρέπεται από τις ε, συνθήκες κρατώντας τα χρήματα στις χώρες τους θα χρειαστεί να τα λάβουμε υπόψη αυτά στην μεταβατική περίοδο. Και μέσα στη μεταβατική περίοδο εντάσσεται βεβαίω και το Brexit, καθώ και η συμπεριφορά τη Μεγάλη Βρετανία απέναντι στον προπολογισμό. Ώστε για τον προπολογισμό του 2020 θα πρέπει να κάνουμε εκεί την προσπάθεια συνδυασμού και με τι προσπάθειε των ε, εισηγητών μα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τα πράγματα εκεί υπόσχονται να είναι αρκετά συναρπαστικά. Αναμένω λοιπόν ε, με χαρά την συνεργασία σας και βεβαίως τις παρατηρήσεις που θα θελήσετε να μου υποβάλλετε. Εξαιρετικά όλα αυτά που μας είπατε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Την κυρία Κλωνεκ Μωρά πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και βεβαίως ε, απευθύνομαι ιδιαίτερο στην εισηγήτρια, αλλά και σε όλους τους υπολείπους. Ε, χαίρομαι πολύ γιατί οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες συνέβαλαν ε, στην προετοιμασία αυτού του προϋπολογισμού. Πρόκειται για τον ε, τελευταίο προϋπολογισμό του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και ε, μάλιστα ε, ιδιαίτερος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές σε αυτή την περίοδο πρέπει να πούμε ότι και μετά από τις ανταλλαγές που είχαμε και τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί στα πλαίσια του Brexit το ενδιαφέρον γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Θα ήθελα βεβαίως να σας ευχαριστώ κυρία Ισηγήτρια για τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές που μας μεταφέρατε σε αυτή την συνθετική βεβαίως ε, εργασία την οποία θα προσπαθήσουμε να ε, εμπλουτίσουμε γιατί αυτή η εργασία σας αποτελεί μια καλή βάση διαπραγμάτευσης για την πολιτική μου ομάδα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Βεβαίως η, ε, έκθεση βασίζεται στις δημοσιονομικές προτάσεις ας το πούμε του Ηνωμένου Βασιλείου και επομένως θα πρέπει λίγο να βάλουμε σε σουρδίνα κατά κάποιο τρόπο τις υποσχέσεις. Ε, πάντως ε, ο προπολογισμό ε, είναι και πρέπει να είναι φιλόδοξος. Αποτελεί όπως είπατε και εσείς γέφυρα προ το επόμενο πι και πραγματικά δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό ότι δηλαδή προετοιμάζεις όσον αφορά ε, προετοιμάζει μάλλον για το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27. Επίσης ε, έχει στόχο να αποφευχθεί κρίση πληρωμών που έχουμε ήδη αντιμετωπίσει και να προβλέψει μια νέα κρίση πληρωμών το 2020 και κυρίως για θέματα όπως είναι η πολιτική συνοχής Επομένως είναι πολύ θετικό που προβλέπονται λύσεις. Επίσης ε, ε, χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ευελιξίας που ε, παρέχει το ΠΙΔΕΛΤΑΠΙ, καθώς επίσης και όλες οι διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποίησαμε ήδη από το 2019 στην προετοιμασία του προϋπολογισμού. Καινοτομία, απασχόληση, έρευνα, πολύ σημαντικά θέματα. Επίση, προωθεί και την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα, υπογραμμίζοντας βεβαίω την ανάγκη ολοκληρωμένη πολιτικής διαχείρισης των εξωτερικών σύνορων και προστασίας τη επικρατεία. της Και εγώ θα ήθελα να τα συνδέσω τα δύο αυτά. Αυξήσει αυξήσεις επίσης όσον αφορά το Erasmus Plus και ε, το σύνολο των εργαλείων που επιτρέπει την καταπολέμηση της ε, νεανικής ανεργίας. Επίσης ε, βοηθούνται οι, όσοι δρούν σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να βοηθηθούν. Επίσης υπάρχει και μια πτυχή ιδιαίτερα σημαντική που αφορά την υποδοχή, την πολιτική υποδοχή, αλλά και την ενσωμάτωση των υποδεχομένων. Ε, Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε αποσαφηνήσει. Εργαζόμαστε όλοι μαζί πάνω σε αυτέ. Πιστεύω ότι η κοινωνική διάσταση του προπολογισμού, του ευρωπαϊκού προπολογισμού, πρέπει να υπογραμμίζεται και ο προπολογισμό του 2020 θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στραμμένο προ τι μελλοντικέ γενναίε. Και εγώ θα ε, κοιτάξω και θα είμαι πολύ προσεκτική όσον αφορά την ε, δράση απασχόληση για του νέου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε αυτή την νέα δημοσιονομική χρονιά, να αντιμετωπίσουμε λέω, το πρόβλημα των νέων που δεν έχουν κατάρτιση και δεν ε, ε, έχουν εργασία. Επίσης, εν ώψη και του επόμενου πιδελταπή θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, υλοποιηθεί και να σχηματοποιηθεί αυτός ο κοινωνικός πολώνας, πυλώνας. Πρόθεση επίσης της κοινωνικής συμπερίληψης και της καταπολέμησης κάθε διάκρισης. Επίσης, σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή θα ήθελα να αναφερθώ ε, στον, στην παρακολούθηση που θα πρέπει να είναι οικονομική, κοινωνική ε, και ψηφιακή. Ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να υποστηρίζει ε, την οικονομία αλλά να είναι στραμμένος προς μια βιώσιμη κοινωνία, πράσινη, ανοιχτή κτλ. Εν συμπεράσματι, να υπενθυμίσω το εξή, το είπα και προηγουμένω: Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα γιατί ε, αυτό είναι άρεκτα συνδεδεμένο με πολιτική προστασία των εξωτερικών σύνορων. Και επίσης συμμερίζομαι κυρία η την, το μέλημά σα για την ασφάλεια των πολιτών. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, διασφαλίσουμε και την προστασία τους, καθώς επίσης και στοιχεία τα οποία άπτονται τη ηθαγενεία τους. Πιστεύω ότι με την ενίσχυση της ασφάλειας θα πρέπει να πούμε ότι ναι, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει αλλά και που προστατεύεται και επομένως η έννοια αυτής της, ε, της ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η πρώτη ανταλλαγή που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Euh, ε, και οπωσδήποτε προσδοκούμε επικοδομητική μελλοντική εργασία, όσο πιο επικοδομητική και καρποφόρα γίνεται να είναι η συνεργασία μας. Ευχαριστώ, Νίλ Στόρβαλς. Έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους ε, ε, για αυτό το έγγραφο το οποίο είναι εξαιρετικό δεν μπορώ να πω περισσότερα στα γερμανικά θα μπορούσα ενδεχομένω να συνεχίσω αλλά δεν είναι και τόσο απλό όταν πρωτοδιάβασα το έγγραφο αυτό Ήταν ευχάριστη η έκπληξη. Ήταν πολύ λίγα τα σημεία στα τα οποία διαφωνούσα. Βεβαίω, αρκεί κανεί να το ξαναδιαβάσει μια δεύτερη, μια τρίτη φορά για να δει κάποια πράγματα που λείπουν. Η κυρία Ολμάιερ είπε και όλοι γνωρίζουμε ότι ε, είναι βεβαίως ε, υπάρχει ένας περιορισμός ε, στο πόσες λέξεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, στο μέγεθος του εγγράφου, Δηλαδή κάποια πράγματα ενδεχομένω λείπουν όχι επειδή δεν ήθελα να το συμπεριλάβει η κυρία Ολμάιερ, αλλά επειδή δεν υπήρχε χώρο. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη, την, τον προπολογισμό που βασίζεται στην απόδοση, το ανέφερε και η Μόνικα. Ε, τα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αυξήσει τον προπολογισμό για την καταπολέμηση του κλίματο και βέβαια στη μάχη δεν έχει κερδιθεί ακόμα. Θέλω να το πω για άλλη μια φορά έτσι ώστε να το θυμηθεί και η Επιτροπή όταν ε, θα σχεδιάσει τον προπολογισμό για το 2020. Καλό θα είναι επίσης ο προπολογισμό να ε, αφορά να είναι ανθεκτικό σε ό,τι αφορά το κλίμα και σε ό,τι αφορά ε, τη βιωσιμότητα. Υπάρχουν όμως και δύο σημεία που είμαι κάπως επιφυλακτικός για την απόδοση. Το εύση πρώτα απ' όλα και η ε, πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων. Και δεν θέλω βεβαίω να μιλήσω κατά ε, της συναδέλφου που μίλησε υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής για την απασχόληση των νέων. Όμως εδώ έχουμε αυτό που ονομάζουμε crowding out. Το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αλλού τέτοιου προγράμματα. Δεν συνάδει δηλαδή με την ε, υποχρέωση προσθετικότητας προσθέμενης αξία Η πρωτοβουλία για την αποσχόληση των νέων θα πρέπει να δώσει μια προστιθέμενη αξία, να μην ε, αντικαταστήσει δηλαδή, τις εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Ε, και εδώ λοιπόν έχουμε αυτή, το φαινόμενο του crowding out, όπως και νωρίτερα, όταν είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση της επιστήμης. Και ξαφνικά είδαμε ότι τα κράτη-μέλη άρχισαν να μειώνουν το δικό τους προϋπολογισμό στους τομείς αυτούς. Πάντα λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος ε, όταν παίρνει μια πρωτοβουλία που φαίνεται πολύ καλή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη-μέλη μετά ε, κάνουν κάτι πολύ κακό, διότι κάνουν περικοπές στους συγκεκριμένους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό πάντα. Υπάρχει μια παράγραφος. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παράγραφος 11. Βεβαίως και πρέπει να εξασφαλίσουμε πολιτική, ε, κοινωνική συνοχή για τους πιο ηλικιωμένους. Στη Φιλανδία μάλιστα υπάρχει ένα σκάνδαλο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την πέθαλψη των ηλικιωμένων και τη φροντίδα. Είναι ένα θέμα σε πολλά κράτη-μέλη, ένα, θέμα έτσι καυτό, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να γνωρίζουμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε των κρατών και τι είδου περίθαλψη θα πρέπει να χρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο και τι σε ευρωπαϊκό. Τώρα, ο καλό μου φίλο ο Ζεράντε πρέπει, μου κάνει κάτι χρήσιμο κάπου αλλού, έτσι ελπίζουμε σίγουρα θα μιλούσε για την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανάγκε των τομέα τη μετανάστευση. Η Μόνικα όμω το ανέφερε ήδη, οπότε νομίζω ότι θα βρεθεί μια καλή λύση. Θα υπάρξει δηλαδή μια καλή συνεργασία μεταξύ των σκληρών εισηγητών και μπορεί τελικά να οδηγηθούμε στην καλύτερη γνωμοδότηση που υπήρξε ποτέ εδώ. Μάλιστα. Υπόσχεσαι πολλά. Τζόρτι Σολέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μόλις συζητήσαμε την αβεβαιότητα σε σχέση με τον προβλησμό του 2019 λόγω του Brexit αλλά η ζωή συνεχίζεται με ή χωρίς Brexit και θα πρέπει βεβαίως ε, να εργαστούμε επί ε, της, ε, του μελλοντικού προπολογισμού Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την, πρόταση και τις κατευθύνες γραμμές. Χαίρομαι καταρχήν που δεν είναι ένα έτσι μακροσκελές έγγραφο με ένα ευχολόγιο. Είναι μια σύντομη περιεκτική πρόταση. Συμφωνώ με πολλά από αυτά ε, τα οποία τονίσατε. Την ανάγκη παραδείγματο χάρη να αποφύγουμε μια κρίση πληρωμών Έχουμε εμπειρία ε, και, από, και στα πρώτα, στις πρώτες χρονιές του παρόντος πολιτικού δημοσιονομικού πλαίσιου όπου αντιμετωπίσαμε μια τέτοια κρίση και χρειάστηκε να βρούμε ένα μηχανισμό για να μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Συμφωνώ επίσης με το γεγονός ότι στο τέλος της έκθεσης αναφέρεστε σε ένα δύσκολο ζήτημα, το άστρο 15.3. Έχουμε εμπειρία από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ε, για τον προβλησμό του 2019 σχετική. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε σαφές το Συμβούλιο ότι χρειάζεται σαφήνεια κατά πόσο το άστρο 15 παράγραφος 3 έχει γίνει κατανοητό πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη και κατά πόσο είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν, να εφαρμόσουν αυτό το άρθρο. Συμφωνώ επίσης με την ανάγκη να προωθήσουμε πιο έντονα την καινοτομία, να δοθεί άμφαση στην ανεργία, στις ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στους νέους και πολλά άλλα. Όμως ο συνήθως προπολογισμό ε, δεν αφορά μόνο αριθμού, αφορά και πολιτικέ προτεραιότητε. Όχι μόνο για τον προπολογισμό του 2020, αλλά για όλη την περίοδο. Όπω γνωρίζετε, η ομάδα μου θεωρεί ότι δεν επικεντρωνόμαστε στι πιο δύσκολε προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ένωση και θα τι δούμε μπροστά μα στο μέλλον. Κλιματική αλλαγή και κοινωνική συνοχή αυτά τα δύο μεγάλα περίπλοκα ζητήματα πρέπει ε, να εξεταστούν πιο προσεκτικά. Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, της κλιματικής αλλαγής είναι ένα θέμα κλειδί για το μέλλον μας. Πρέπει να αποτελεί αυτό οριζόντια προτεραιότητα και αυτό πρέπει να μεταφράζεται και στον προπολογισμό με έναν πιο φιλόδοξο τρόπο από ό,τι τώρα. Πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς μια οικονομία ε, κυκλική, με χαμηλή χρήση άνθρακα έως και μηδενική, ε, διότι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω σχέση με τους στόχους που έχει θέσει για το κλίμα. Ξέρουμε ότι δεν θα επιτευθούν οι στόχοι ε, για το mainstreaming του κλίματος. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στο θέμα αυτό, καθώς και στο θέμα το κοινωνικό, στην κοινωνική διάσταση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθάει για να βελτιωθεί η ζωή αυτών που ζουν δύσκολα στην καθημερινότητά τους και υπάρχουν σχετικά εργαλεία στον προπολογισμό γι' αυτό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Επίσης, ε, διαπιστώνω ότι εδώ υπάρχει μια διασύνδεση έτσι κάπως πονηρή στην έκθεσή σας μεταξύ ασφάλειας και μετανάστευσης ε, πρέπει να έχουμε παρακαλώ την ευρύτερη εικόνα να μιλάμε περισσότερο για την ασφάλεια των ανθρώπων βεβαίως ε, συνοριοφύλακες συνοριοφυλακή, ακτοφυλακή προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτά αλλά το συνδέουμε αυτό με, απλά με την ασφάλεια, μετανάστευση και ασφάλεια δηλαδή, ε, ε, δεν είναι ο πλέον κατάλληλο τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο ζήτημα. Πάντως αναμένω με ανεπιμονησία τη συνεργασία μας για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Νιριάννα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πόσο σύντομη είναι αυτή η γνωμοδότηση. Θα είμαι και εγώ σύντομη στην παρέμβασή μου. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα α, έχουν. Και το Brexit βεβαίως επισκιάζει τα πάντα, αλλά εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Ε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους συμπολίτε μας. Ταυτόχρονα ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ποιος είναι ο αντίκτυπος του Brexit, διότι θα έχει αντίκτυπο στον προπολογισμό. Είναι περίπλοκο λοιπόν. Πρέπει όμως εμείς να εργαστούμε με βάση αυτά που ξέρουμε, όχι με αυτά που μπορεί να συμβούν, αυτά που μπορεί να πούν ή να κάνουν οι Βρετανοί. Πρέπει να έχουμε απτά στοιχεία. Είναι παρεφαρήσεις προτεραιότητες σε πολλούς τομείς, κοινωνική συνοχή, απασχόληση των νέων και σχετική πρωτοβουλία. Καλή πρωτοβουλία αυτή. Βεβαίω υπάρχουν προβλήματα σε κάποιε χώρε όπω η Ιρλανδία. Έχουμε ε, πολύ κακό ε, έτσι, ιστορικό στην απορρόφηση. Ε, το Εράσμους επίση, βεβαίω, Ανησυχώ όμω ότι γίνεται κάπως ελιτιστικό το Εράσμους. Έτσι αφορά μόνο παιδιά τα οποία μπορούν να πληρώσουν ε, ένα σημαντικό ποσό αρχικά, μπορούν να πάρουν ένα δάνειο, ε, Βεβαίω, εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα ε, τη Δημοσιονομική Επιτροπή, είναι πιο πολύ τη Επιτροπή Παιδεία. Το ίδιο ισχύει για ε, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Χαίρομαι που υπάρχει μια αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι, και οι αλληλεί μα. Ε, το βλέπουμε, προσπαθούμε να δούμε πώ στα πλαίσια του e ε, να ε, ισοσκελίσουμε κάπως τα πράγματα. Ε, δεν συμφωνώ τόσο ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σολέ για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Ε, εμείς είμαστε υπέρ της ουδετερότητας. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε ένα, μια, ένα, ένα δρόμο προστατευτισμού. Υπάρχουν όλες άλλες προτεραιότητες, ε, πιο ανθρωπιστικές τουλάχιστον για μας και όχι να μην γίνουμε ένα φρούριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί έχουμε όλοι προσπογράψει ε, να συμμετάσχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπόριο, ειρήνη, ε, ευημερία και όχι ένα φρούριο εάν δουν οι πολίτες ότι εμείς δίνουμε έμφαση στην άμυνα, τη στρατιωτική, περισσότερο από την γεωργική πολιτική, ας πούμε, ή από το να θρέψουμε τους πολίτες μας, ε, εμείς δεν συμφωνούμε. Ε, πρέπει να υπάρχει ευελιξία ε, να επαναξιολογήσουμε αυτά τα προγράμματα καθώς περνάει ο καιρός. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε άκαμπτοι με βάση τις συνθήκες της τωρινές, με το Brexit, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για να επαναξιολογήσουμε αυτά τα προγράμματα ε, όπου χρειάζεται ε, δηλαδή κάποια προγράμματα που θα χρειαστούν υποστήριξη, κάποια, άλλη, ε, κάποια άλλα λιγότερα, ανάλογα και θα γίνει με το Brexit, εφόσον υπάρξει Brexit. Αυτά ε, αναμένω τη συνεργασία μας. Υπομονησία. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τη γενική μας εισηγήτρια. Σας συγχαίρω λοιπόν κύριε Χολμάγερ. Ξεκίνησε λοιπόν μία συζήτηση η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. Θα ήθελα και εγώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, μία πρώτη, σε σχέση με την παράγραφό σας για την έρευνα και την καινοτομία προετοιμασία του μέλλοντος η υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Ε, εάν θέλουμε να εκδημοκρατήσουμε το πρόγραμμα έρασμο, Έρασμος το οποίο αφορά κυρίως τους φοιτητές τώρα, ε, όμως εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει και οι μαθητευόμενοι να έχουν την δυνατότητα ε, να κάνουν αυτό το πρόγραμμα Έρασμους. Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες και οργανισμοί για την μαθητεία. Επομένως, ενδεχομένως ε, ίσως ε, μέσω ε, πιστώσεων συνοχής να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την δυνατότητα μαθητείας σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί η επαγγελματική Συγγνώμη, εάν δώσουμε μια επαγγελματική σωστή κατάρτιση στους νέους, τότε πραγματικά θα υποστηριχθεί και η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Δεύτερη παρατήρηση. Έχω την εντύπωση μάλλον όχι, την προηγούμενη Παρασκευή ε, στο Κανταράς ε, ε, επισκέφτηκα το, την εγκατάσταση ΙΤΕΡ. Δεν μιλάμε πολύ για το ΙΤΕΡ. Η τεχνολογία σχάσης σύνδεξης είναι πολύ σημαντική και είναι συνδυασμένη και με την πυρηνική σχάση. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε κάθε λόγο σαν Ευρώπη να είμαστε περήφανοι. Η Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Κορέα κάνουν ε, επίσης ε, τέτοιες δραστηριότητες, αλλά ε, υπερέχει η Ευρώπη. Εάν μπορέσουμε μέχρι το 2042 να αντισταθμίσουμε ε, την ε, ε, λήξη χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Εάν καταφέρουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες που μέχρι τώρα τα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν και αν από το 1 δις μπορέσουμε να περάσουμε στα 10 δις από εναλλακτικές μορφές ενέργειας ε, τότε θα, θα είναι κάτι σημαντικό και αν μπορέσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να ε, εξισορροπήσουμε τα 150 χρόνια χρήσης των ορυκτών καυσίμων αυτό πραγματικά σημαίνει ότι δημιουργούμε ένα μέλλον που προστατεύει ε, και συμμετέχουμε σε ένα παγκόσμιας εμβέλειας πρόγραμμα και πραγματικά εδώ μπορώ να συμμεριστώ την ελπίδα που έχει και η συγγήτρια. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Μόνικα Χολμάγερ ε, για να κάνει τα τελευταία της, ε, τελευταίες παρατηρήσεις, αλλά να ζητήσω πρώτα τον κύριο Πρεζά, ο οποίος ε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας κάνει τα σχόλιά του. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να στεφθεί από πλήρη επιτυχία η προσπάθεια που γίνεται για τον προϋπολογισμό του 2020. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ε, χαιρετίζω και την ε, έκθεση της εισηγήτριας και την, τα όσα ακούστηκα στην ανταλλαγή απόψεων. Ε, κατανοούμε όλοι βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός σύγκληση σχετικά με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα ε, και βεβαίως και για τις ε, προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των ε, προγραμμάτων ε, γιατί πραγματικά ο αντίκτυπος ε, είναι πάρα πολύ μεγάλος κυρίως όσον αφορά τις πληρωμές γιατί θα συμφωνήσετε όλοι ότι θέλουμε να αποφύγουμε την δυσχερή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε την προηγούμενη φορά. Η υλοποίηση του 2018 είναι μάλλον καθησυχαστική όσον αφορά ε, αυτό το θέμα και επομένως ε, ε, νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε οποιασδήποτε περιπλοκές όσον αφορά το 2020 γιατί νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει υπό καλύτερο έλεγχο το επόμενο ΠΔΠ. Βεβαίως το καλό σενάριο είναι ότι θα υπάρξει συμφωνία εν τέλει με το Ηνωμένο Βασίλειο. και ότι θα υπάρξει μια σταθερότητα. Εάν όμως αυτό δεν ε, γίνει πραγματικότητα, ναι, θα πρέπει να ληφθούν κάποιες ε, διορθωτικές ε, κινήσεις, όπως άλλωστε ανέφερε και ο Επιτροπός κ. Σέτιγκερ το πρωί. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, είναι γνωστό. Στον τριμερή διάλογο θα έχουμε και συζήτηση πλήρους αναλύσεως όλων των στοιχείων και περαιτέρω πρόθεση στο κατευθυντηρίο γραμμών. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική ε, συζήτηση μεταξύ των αρχών του προϋπολογισμού έτσι ώστε να προετοιμαστεί σωστά ε, και το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρέζα, κυρία Χολμάγερ. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ επίσης πολύ όλους τους ε, σκιώδης καθώς και συναδέλφους για τις διάφορες προτάσεις που έθεσαν υπόψη μου και βεβαίω για την συζήτηση. Είτε πρόκειται για θέματα κοινωνικά, όπως είπε ε, προηγουμένως άλλος συνάδελφος, θεωρώ ότι θα πρέπει να καθίσουμε να συνεννοηθούμε ότι επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα δημοσιονομικά θέματα. Για τα υπόλοιπα, εάν δηλαδή προσπαθήσουμε να μπούμε στα επιμέρους ειδικά προγράμματα, θα αντιμετωπίσουμε δυσχέρειες. Το ίδιο για τον έρασμο και άλλα δυστυχώ δυστυχώς καμιά φορά πρέπει να σταθεί κανεί στον πειρασμό να εντάξει, να, συ, ε, εγγράψει και άλλα πράγματα στο κείμενο. Περιορίστηκα στα δημοσιονομικά, ώστε να μην ε, διευρυνθεί υπερβολικά το κείμενο. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Για το θέμα γέι, ο Τόρβαλς έχει δίκιο. Από την άλλη μεριά, από την μια μεριά μάλλον είναι θέμα ειδικό, ειδικού ενδιαφέροντο για μα. από την άλλη μεριά διαπιστώσαμε τι τελευταίες χρονιές με τα ελλείμματα ότι έχει παραγάγει όχι μόνο ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και για προσωρινά μέτρα και αυτό επικρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα, για άλλα θέματα, όπω είπε ο κ. Σαρτούγι, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τι νέε και του νέου, ίσω πρέπει να λάβουμε υπόψη και για παράδειγμα, την δι, διτή κατάρτιση, δηλαδή και την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε μακροπρόθεσμα υπάρχουν ωφέλη για τους νέους και κυρίως να μην υπάρχει μονάχα ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα απασχόλησης ή βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα κατάρτισης που αντί να προσφέρει λύσεις στην πραγματικότητα των νέων δηλαδή, ε, για το μέλλον των νέων, απλώς τους προσφέρει μια σύντομη προσωρινή απασχόληση. Για τα άλλα συμφωνώ. Για το θέμα το μεταναστευτικό, ασφαλώς ε, το έχω περιλάβει ε, εν συντομία, θα το συζητήσουμε βεβαίως και θα χρειαστεί να τοποθετηθούμε. Το ίδιο και για τις συνθήκες που διαβιούν τα παιδιά, κυρίως σε περιφέρειες οι οποίες ε, είναι περιφέρειες συνοχής και εκεί να δώσουμε κονδύλια και σε προγράμματα, έργα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση των μικρών παιδιών και όχι μόνο χρήματα για κατασκευή δρόμων κλπ. Είναι σημαντικό αυτό για τη διαμόρφωση της ζωής τους των παιδιών αυτών. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Εάν τώρα μου επιτρέπετε να πω κάτι για το 15-3. υπάρχει συμφωνία, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κοινοποιήσει ποιες, ποιοι είναι οι όροι υπό τους οποίους θα λαμβάνει η χώρα στο μέλλον το 15-3. Να έχουμε απλώς μια παράγραφο καινού, καινή περιεχομένου δεν μας εξυπηρετήσει τίποτα. Αυτό μας ενόχλησε πολύ άλλωστε και στις συζητήσει για τον προπολογισμό. Θα πρέπει να κάνουμε από κοινού, να υποβάλουμε από κοινού το αίτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξεκαθαρίσει δηλαδή τους όρους υπό του οποίους θα λειτουργήσει το 15-3. Κάτι το οποίο δεν έχει σημειώσει τώρα. Έχω και δύο ερωτήσει Αφενό το ITER, υπάρχουν και τεχνολογίες που δεν είναι καν γνωστές στο κοινό, εκτός από την σύνδεξη τώρα, σε ό,τι αφορά την βελτιωμένη χρήση της ενέργειας. Για παράδειγμα, για την χρήση κινητών και την χρήση νέων ε, τεχνολογιών για την αυτόνομη ε, φόρτιση του κινητού και ούτε καθεξής. Όντως από την άλλη μεριά το ίτερ δεν λαμβάνει επαρκή προσοχή και με τους ε, λογαριασμούς του θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα από το 2020 και μετά. Διότι προχωρούν με το έργο αυτό, το ίτερ δηλαδή, τη σύνδεξη, και εμείς δεν το έχουμε λάβει επαρκώς σοβαρά υπόψη αυτό για να προβλέπουμε τη σχετική χρηματοδότηση. Και τώρα ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσω με του και οδησυγητές και συγκήτριες, όπου δεν είμαι βεβαία πώ θα το αντιμετωπίσουμε, έχουμε τη συζήτηση δηλαδή περί ιδίων πόρων από την φορολόγηση ψηφιακών ομίλων επιχειρήσεων. Θα το συζητήσουμε αυτόνομα ω θέμα ή θα το εντάξουμε στο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλω να γνωρίζω τη γνώμη σα, διότι έχει μεγάλη σημασία για τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Δεν είμαι βέβαια αν πρέπει να το βάλουμε ήδη στο προπολογισμό του 2020 ή αν πρέπει να περιοριστούμε στη συζήτηση για το ΠΔΠ. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, γιατί δεν είμαι βέβαια, ξαναλέω, αν πρέπει να μπει στον προπολογισμό του 2020 μέσα στα πλαίσια της μετάβασης προς το ΠΔΠ. Τέλος, Brexit. Για το Brexit, το κέριο ερώτημα για μένα, για το 2020 δηλαδή, είναι είναι εάν θα παραβεί τις συνθήκες η Μεγάλη Βρετανία, διότι έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό μέχρι τέλος 2019, αρχής 2020. Και ακούμε και το ενδεχόμενο να μην ε, σεβαστεί τις ε, υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη μέχρι το 2020. Τώρα, οι βασικέ συνέπειε, εφόσον, δεν, εφόσον παραβεί τι υποχρεώσει τη Μεγάλη Βρετανία, οι μεγάλε συνέπειε θα αρχίσουν πια από το 2021. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή γραμμή. Ευχαριστώ κυρία Συγήτρια, κυρία Γενική Συγήτρια. Είναι αλήθεια ότι σε σχέση με το Brexit έχουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει σε όλες τις φάσεις διαπραγματεύση και ότι δεν συνέβη το ίδιο με το Westminster. Ίσως ε, μάλιστα αυτό να κάνει και τη διαφορά. Λοιπόν, θα είμαστε σύντομοι σε ό,τι αφορά ψηφοφορίες. Ψηφοφορίες δεν υπάρχουν. Να σας πω όμως για το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση της κυρίας Ολμέγερ 14 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι ε, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στην έκθεση της κυρίας Ολμέιερ. Θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τις τροπολογίες της 26 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή τη Δημοσιονομική θα λάβει χώρα 7 Μαρτίου έτσι ώστε να ψηφιστεί στη συνέχεια σε κάποια ψολομέρεια στο Μαρτίου το χρονοδιάγραμμα βεβαίως ε, ε, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με τον κύριο Έτιγκερ ε, θα ήταν καλό η θητεία του να συνεχιστεί μέχρι 30 Νοεμβρίου για να συμβεί κάτι τέτοιο αλλά δεν νομίζω να μπορεί να γίνει αυτό πάντως σίγουρα θα διευκόλυνε το συντονισμό και την συνέχεια Λοιπόν, αυτά για τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ε, κάτι, κάτι ενημερωτικό ούτε για τα στεγαστικά. Λοιπόν, 14 Φεβρουαρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Θα εξετάσουμε ένα σχέδιο τότε ε, σχετικά με τα κίνητα και θα ακούσουμε και για το Γενικό Γραμματέα και την έκθεσή του και το σχέδιο του προπολογισμού του, του Κοινοβουλίου μάλλον το 2020. Δηλαδή ταυτόχρονα το Προεδρείο και η έκθεση της Γραμματείας ε, θα ενημερώσει ε, την Επιτροπή Προπολογισμού. Είναι σημαντική η πρόοδος αυτή, να ενημερωθούμε ταυτόχρονα. Στις 18 Φεβρουαρίου, πολύ σημαντική εβδομάδα, διακοινοβουλευτική, οπότε παρακαλώ να είστε εδώ, διότι θα έχουμε έτσι μια αρκετά έντονη ε, έτσι, ανταλλαγή απόψεων με τους ε, συναδελφούς μας εθνικούς βουλευτές και 26-27 Φεβρουαρίου Επιτροπή Δημοσιονομική θέλει κάποιο το λόγο υπό τα διάφορα, κανείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας πέρα στη συνεδρίαση.